λάβαμε ε, μία αίτηση σε σχέση με διορισμούς σε ε, αντιπροσωπείες και έχουν εγγραφεί στα πρακτικά. Ε, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θεωρούμε ότι εγκρίνονται.